περίοδο που ήταν αφηρημένη στι μονόλεπτε παρεμβάσει, πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση πριν να κλείσουμε την απόψινή σύνοδο και αυτή αφορά την ομάδα Γκουε, από την οποία έχω λάβει ένα αίτημα, ότι ο κύριος Γιαρομίρη Κόλιτσεκ να διοριστεί ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, Σύνδεσης με την Ουκρανία, Ένωση Ουκρανία. Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, γκρίνεται αυτός ο διορισμός και η επόμενη